που με βοήθησαν σε αυτό το πολύ πολύπλοκο και δύσκολο έργο, αξιόλογο όμως σε τελευταία αναλύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ντεμπρόν και όσους συναδέλφους μίλησα. Έληξε η συζήτηση ή ψηφίζουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι για αυτό το θέμα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της οδηγίας για το πακέτο ταξιδίου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αξιότιμα μέλη, χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία για να σας ενημερώσω σε σχέση με την αναθεώρηση του πακέτου ταξιδίων. Όταν εγκρίθηκε αυτή η οδηγία το 1999, τα πακέτα αυτά τα ταξιδιωτικά ήταν πάρα πολύ συνηθι. Από τότε η αγορά έχει μεταβληθεί σημαντικά. Η εξέλιξη του ίντερνετ δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ναι, κάνουν τις κρατήσεις τους απευθείας στα ξενοδοχεία και στις αεροπορικές εταιρείες. Έχει ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Οι περισσότεροι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα οργανώνουν μόνοι τους τις, αλλαγές, τις διακοπές τους αντί να αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται καλύτερα οι καταναλωτές όταν πηγαίνουν διακοπές. Ξέρουμε επίσης ότι η οδηγία αυτή έχει δημιουργήσει άνισο περιβάλλον για τους πράκτορες και ορισμένοι ε, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις αν και πουλούν παρόμοια προϊόντα. Η ελάχιστη εναρμόνιση έχει φέρει και νομικό κατακαιρματισμό στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή νομοθεσία μπορεί να μην είναι επικαιροποιημένη. Γι' αυτό κάναμε ε, προχωράμε σε μία αξιολόγηση της κατάστασης για να συνεχίσουμε μετά στην αναθεώρηση ε, των διατάξεων για τα οργανωμένα ταξίδια. Ε, δημοσιεύσαμε ακόμη μία έκθεση όσον αφορά τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές από τα αποκαλούμενα δυναμικά πακέτα. Ξεκινήσαμε και μία δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας και έληξε αυτή η διαβούλευση στις 7 Φεβρουαρίου. Η Κομισιόν τώρα εξετάζει πάνω από 100 παρατηρήσεις τις οποίες θα περιλάβει στην αξιολόγηση και το εύρος της αναθεώρησης θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Θα σας πω όμως ποιες είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Πρώτον, θέλουμε υψηλό επίπεδο προστασίας. Είναι το κλειδί αυτό, αν θέλουμε να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές όταν αγοράζουν διακοπές. Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα ταξίδια, εφόσον οι διασυνοριακές αγορές είναι συχνές σε αυτό το τομέα. Συνεπώς χρειάζεται περισσότερη εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Τέλος, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες για τους πράκτορους που πουλούν οργανωμένα ταξίδια. Η Κομισιόν πιστεύει ότι θα υποβάλει τις προτάσεις αρχές του 2011 και η πρόκληση είναι να προσδιορίσουμε σωστά το εύρος της οδηγίας η Κομισιόν θα εξετάσει τις δυνατότητες απέκτασης της οδηγίας ώστε να καλυφθούν περισσότερες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις ακόμη και αυτά τα δυναμικά πακέτα όπως αποκαλούνται. Αυτό θα προστατεύσει καλύτερα τους καταναλωτές να πηγαίνουν διακοπές. Πρέπει ακόμη να επικαιροποιήσουμε τις προϋποθέσεις ενημέρωσης και την αστική ευθύνη των μερών στη σύμβαση αυτή. Ακόμη, για να ενισχύσουμε την συνειδητοποίηση των καταναλωτών, θα εισαγάγουμε ένα τυποποιημένο πακέτο ρυθμίσεων για οργανωμένα ταξίδια. Ακόμη, θέλουμε να ενισχύσουμε την προστασία κατά της πτώχευσης πρακτόρων, όπως άλλωστε αυτό μας ζητήθηκε πρόσφατα και από το Ευρωκοινοβούλιο. Στην αρχή του 2009 ε, δημοσιεύσαμε μία ανεξάρτητη μελέτη που εξέτασε τις διάφορες δυνατότητες αντιμετώπισης των πτωχεύσεων. Επίσης, εξετάζουμε τα δικαιώματα των επιβατών περαιτέρω για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε την καλύτερη προστασία κατά των πτωχεύσεων στο Ευρωκοινοβούλιο πριν από το τέλος του 2010. Ευχαριστούμε. Πρώτος ομιλητής ο κύριος Σουάμπ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ντάλη για την υποστήριξή του ώστε να γίνει αυτή η τροποποίηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι και έγκαιρη αυτή η τροποποίηση γιατί θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στις διακοπές της Πεντηκοστής και επέκεινα. Υπάρχουν ήδη μια σειρά από θέματα τα οποία τίθενται σε ό,τι αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και που θα πρέπει να τροποποιηθούν για να υπάρχει καλύτερη τροποποίηση των καταναλωτών σε σχέση με τα δικαιώματά τους. Σήμερα έχουμε πολλές πλατφόρμες στο ίντερνετ οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα με περαιτέρω συνδέσμους να κλείσουν περαιτέρω κρατήσεις ταξιδιωτικές οι καταναλωτές παρά το γεγονός ότι αυτές οι κρατήσεις οι πρόσθετες δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. Οι φτηνές αυτές λοιπόν πτήσεις, γιατί για αυτές κυρίως ε, πρόκειται, δεν υπόκεινται στις ε, ε, ανάγκε πληροφόρηση των καταναλωτών που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη-μέλη και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη δυνατότητα του καταναλωτή να τύχει τι κατάλληλη πληροφόρηση και να μπορέσει να ε, εγείρει και να εκμεταλλευτεί τα δικαιώματά του. Επίση, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του κατά πόσο τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών πτήσεων θα πρέπει να καλύπτονται μαζί με τα δικαιώματα των ε, πελατών των οργανωμένων ταξιδίων σε ένα κοινό έγγραφο το οποίο θα έχει το νομοθετικό χαρακτήρα και θα καλύψει όλο αυτό το πεδίο του επιστητού. Τρίτον, κύριε Επίτροπε, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τα γραφεία ταξιδίων. Αυτό δημιουργεί προβλήματα βέβαια σε ό,τι αφορά τα διαμεθοριακά ταξίδια. Σε ορισμένες χώρες αναφέρονται ως γραφεία οργανωμένων ταξιδίων, ενώ στη δική μου χώρα έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Αυτό οδηγεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα όταν θέλουμε εμείς να έχουμε τουλάχιστον μια βασική συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ταξίδια και τις ενέργειες αυτών των γραφείων που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Τέλος, πιστεύω ότι χάρη στο ίντερνετ και μια περισσότερη χρήση <clears throat> του ίντερνετ θα πρέπει ο καταναλωτής να γνωρίζει ποιε είναι οι δυνατότητε κλεισίματο από το Ιντερνετ, αλλά παράλληλα να έχει την κατάλληλη πληροφόρηση και να αποφευθούν οι καταχρήσει. Ο κύριο Κέλλη. Για δύο λεπτά. Ολόκληρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση αυτή γίνεται σε πολύ καλή στιγμή. η συζήτηση για το μέλλον του τουρισμού και των αεροπορικών μεταφορών, δηλαδή, μετά από τα προβλήματα που γνωρίσαμε εγκατάλειψης ταξιδιωτών διότι επτόχευσαν ορισμένες χαμηλού κόστους εταιρείες ιδιαίτερα. Ξέρουμε πολλές περιπτώσεις ταξιδιωτών που αφέθηκαν μόνοι στην τύχη τους χωρίς καμία πληροφόρηση και χωρίς καμία δυνατότητα να μάθουν τι πρόκειτο να τους συμβεί. Γι' αυτό είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση και πρέπει η Κομισιόν να λύσει αυτό το πρόβλημα γιατί το έχουμε αφήσει εκρεμές πολύ καιρό. Πριν από 10 χρόνια υπήρξαν άλλες οδηγίες, ταξιδιωτικές οδηγίες για να τις πω έτσι, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες μεταξύ κρατών είναι κάτι που πρέπει να διευθετηθεί περαιτέρω. Ήδη όμως οι προτάσεις είναι απαρχαιωμένες. Δεν χρησιμοποιούν οι καταναλωτές πια τόσο πολύ τα οργανωμένα ταξίδια. Το 40% στην Ιρλανδία αυτοοργανώνονται. Οι περισσότεροι μόνοι τους κάνουν τις κρατήσεις. Είναι σαν να είναι ο καθένας ταξιδιωτικό γραφείο από μόνος του. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να δείξουμε εδώ είναι να δείξουμε ότι ο καταναλωτής, να δείξουμε στον καταναλωτή ποιος είναι υπεύθυνο κάθε φορά για κάθε πρόβλημα. Να έχει σαφέστατη πληροφόρηση. Να πληροφορείται ο καταναλωτής αλλά και η καταναλώτρια. Παρακαλώ κύριε Κέλλη, λέει ο πρόεδρος, μπορείτε να μιλάτε πιο αργά γιατί οι ερμηνευτές και οι ερμηνεύτριες δυσκολεύονται. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σαφείς ευθύνες. Ποιος ευθύνεται όταν γίνει, συμβεί κάτι, το ταξιδιωτικό γραφείο, η αεροπορική εταιρεία, κανείς δεν το ξέρει. Κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς σε ποιον να απευθυνθεί. Πρέπει η ευρωπαϊκή οικονομία που ήδη βασίζεται σε διαμεθοριακές συναλλαγές να διευθετηθεί, να τύχει διευθέτηση και για τα ταξίδια. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να βρει κανείς ποιο είναι το τμήμα παραπώνων μιας αεροπορικής εταιρείας άρα αυτό που ζητάμε είναι ακόμη πιο δύσκολο να υπάρχει τμήμα παραπώνων και για, τις αεροπο... και για τα ταξίδια, για τα ε, πρακτορία. Πρέπει η νομοθεσία αυτή όχι απλώς να ενημερωθεί αλλά να δημιουργηθεί νέα νομοθεσία. Τέλος, κάτι που μπορεί να το σκεφτεί η Κομισιόν είναι πόσο στοιχίζει μια πτήση. Όλοι ξέρουμε ότι οι τιμές που αναφέρουν οι διαφημίσεις δεν συμπεριλαμβάνουν φόρους ε, και άλλα έκτακτα έξοδα όπως πρόσθετες αποσκευές κλπ. Δεν, είναι, λοιπόν, δεν υπάρχει μεγάλη διαφάνεια στην διαφημιστική πληροφόρηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε θα ήθελα εξ ονόματο τη ομάδα των Φιλελευθέρων να χαιρετήσω την παρουσία σας και να σε ευχαριστήσω και να τονίσω ότι είναι σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση της οδηγίας. Πράγματι, κυρίε και κύριοι, μπορούμε να χαιρόμαστε ότι ζούμε στην Ευρώπη και ότι μπορεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί κανείς να συζητά θέματα όπως το πώς ταξιδεύει κανείς σε οργανωμένα ταξίδια μαζί με τα ζώα του. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν οι απαραίτητε ρυθμίσει για την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των ζώων. Αλλά το βασικό δικαίωμα των καταναλωτών για ταξίδια στην Ευρώπη, η ελευθερία διακίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει εμεί να την εξασφαλίσουμε. Πριν από 20 χρόνια είχαμε περάσει αυτή την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια πριν από, για να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που θέλει να γνωρίσει ο πολίτη στην ομορφιά και άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να γίνεται αυτό με πλήρη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Να μην συμβεί λοιπόν κάτι το οποίο δεν θα λειτουργήσει κακό, άσχημα χωρί να υπάρχει δυνατότητα αποζημίωση. Ο κύριος Επίτροπο τονίζει ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην ε, οδηγία, αλλά εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε την προσοχή του ότι υπάρχουν ακόμα κενά στο συστήμα, γιατί πάρα πολλοί καταναλωτέ κλείνουν μόνοι του, όχι από γραφεία, αλλά μέσα από το ίντερνετ τα ταξίδια του και είχαμε θέσει και ένα ερώτημα ως Επιτροπή Μεταφορών διότι υπήρξαν προβλήματα παγκοσχά στην Σλοβακία όταν ε, εταιρείε χαμηλού κόστους τους είχαν αφήσει χωρίς κανένα, καμία αποζημίωση, χωρίς καμία δυνατότητα να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Έχουμε επικρίνει όλοι τις, φτω, τις πτήσεις και τις εταιρείε που λειτουργούν στο ίντερνετ με αυτόν τον τρόπο. Θέλουμε να υπάρχει όμω η χρήση αυτών των κτηνοπτήσεων, αλλά με τρόπο που θα εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι ελλείψει σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, πώ θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά. Αυτό κάνει απαραίτητη μια τροποποίηση αυτή τη οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια και θα πρέπει να δούμε αν χρειάζονται περαιτέρω να γίνουν ενέργειες όπως είπε και ο συνάδελφός μου προηγουμένως, συγκεκριμένες ενέργειες και τροποποιήσεις για τα αεροπορικά ταξίδια. Είναι χρήσιμο λοιπόν να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα και εγώ προσβλέπω στο να αντιμετωπίσουμε όχι φυσικά μόνο τα θέματα των ζώων, τα οποία είναι και αυτά σημαντικά, αλλά κυρίως των καταναλωτών και των επιβατών των αεροπορικών πτήσεων στην Ευρώπη, για να έχουν πλήρη ε, κάλυψη των δικαιωμάτων τους. Κυρία Μπρέκου, για λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Βρισκόμαστε τώρα σε ένα πλαίσιο το οποίο μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των ε, ταξιδιωτών. Αλλά και οι εταιρείε ε, οι οποίες παρέχουν ε, οι υπηρεσίε στον τομέα των οργανωμένων ταξιδίων θέλουν και αυτέ να εξασφαλίσουν να γίνεται με τον πιο ομαλό δυνατό τρόπο αυτό το, αυτή η ενέργεια. Παρά το γεγονό ότι έχουμε περισσότερου ταξιδιώτε συνέχεια, έχει μειωθεί ο αριθμό των ατόμων που καλύπτονται πλέον από την ευέλευτη τη οδηγία και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διεκδικήσει την ανάγκη να υπάρξει μια επανεπεξεργασία αυτή τη ε, οδηγία. Έχει κλείσει ο γύρος διαφολεύσεων και έχουμε φτάσει πια στο σημείο που θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις. Εγώ χαιρετίζω τη δήλωση του κυρίου Νταλή. Αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα ήθελα και πάλι να απευθυνθώ στον Επίτροπο. Καταρχήν, ο τομέας εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να είναι ευρύτερη και αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες μόνοι τους καταρτίζουν ένα πακέτο ταξιδιωτικό και αυτό χρησιμοποιώντας το διαδικτύο. Έχουμε δει όμω ότι πολλέ φορέ υπάρχουν προβλήματα, Όπω με το Eurostar, όπου εκατοντάδε χιλιάδε σχεδόν τουρίστε αντιμετωπίσαν προβλήματα, δεν πήραν καμία αποζημίωση. Δεν υπήρξε η δυνατότητα αποζημιώση για, για την απώλεια των ε, κρατήσεών του σε ξενοδοχεία από το γεγονό ότι χάσανε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν θεατρικέ παραστάσει στο Λονδίνο, παραδείγματο χάρη. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μια νέα ρύθμιση. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις στα κράτη-μέλη και υπάρχει και διαφορετική φυσικά συμπεριφορά των, ε, των ταξιδιωτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Ακόμα και η αντίστοιχη νομολογία είναι ποικίλη. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που μας κάνουν απαραίτητη μια τροποποίηση της οδηγίας. Δεν είναι επίσης πολλά θέματα σαφή. Τι ακριβώς είναι ένας μεσίτης ταξιδίων, ένα πρακτορείο ταξιδίων. Τι σημαίνει επίσης ανώτερη βία όταν υπάρξει μια ακύρωση. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να προχωρήσουμε σε κάποιες ρυθμίσεις ώστε ο τομέας των ταξιδίων να μπορεί να έχει μια σαφήνεια. Έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε που πήραμε μετά από τι διαβουλεύσει μα με του εμπλεκόμενου και με, μου, με, μου δίνει ακόμα μεγάλη εντύπωση ότι δεν έχουμε καταλήξει σε μια, σε μια απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε μία σαφήνεια στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο αλλά και στην ευθύνη που έχουν οι πράκτορες ταξιδίων, ο οποίος θα πρέπει να διασαφινιστεί καλύτερα, γιατί όλο και περισσότερο κατακλείζονται οι ταξιδιώτες με πληροφορίες από το ίντερνετ, αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι πάντα ακριβής ή χρήσιμη. Πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν παραπλανητικές πληροφορίες, όπως πραγματικά τους λένε ότι θα πρέπει να πληρώσουν κάποιες επιβαρύνσεις για κατοικίες τις οποίες νοικιάζουν, οι οποίες είναι ανύπαρκτες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει προστασία και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει πτώχευση των ταξιδιωτικών γραφείων. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει προστασία. Ξέρω ότι στην περίπτωση των κάτω χωρών μεταξύ Φλάνδρας και Ολλανδίας υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες οι οποίες υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Είναι πολύ εύκολο να υπάρξει η σύναψη μια σύμβαση σε ένα κράτος, αλλά να εκτελεστεί η σύμβαση σε ένα άλλο κράτος μέλος. Επίσης, το θέμα των τιμολογίων. Υπάρχουν στα περισσότερα κράτη οι λεγόμενες all-inclusive τιμές, οι περιεκτικές τιμές οι οποίες παραλαμβάνουν τα πάντα. Ε, <clears throat> τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Επιπλέον, πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η έννοια ανωτέρα βία. Είναι απαραίτητο να υπάρξει και μία υποχρέωση παροχή πληροφοριών σε σχέση με το τι αποτελεί ανώτερη βία. Και επίση να υπάρχουν οι αντίστοιχε κυρώσει σε περίπτωση παραβάσεων. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα όπω πρέπει. Ο κύριος Μπίλεν, δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κοινοτική οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια που συζητούμε σήμερα ανατρέχει στο 1990, πριν 20 χρόνια. Τότε ήταν η εποχή όπου η πιο δημοφιλής ε, μορφή ταξιδιού ήταν ε, δύο εβδομάδες ταξίδια οργανωμένο μέσω ε, πρακτορείου και με τη βοήθεια ενός καταλόγου. Η οδηγία αυτή τώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει με μέτρα προστασίας τα ζητήματα που αφορούν τον καταναλωτή, ζητά διαφάνεια, επιτρέπει τη δυνατότητα διακοπής οποιασδήποτε εμπορική σχέση με το πρακτορείο και προστασία του ταξιδιώτη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια άλλαξε ριζικά και τελείως το επιχειρηματικό μοντέλο αλλά και το καταναλωτικό μοντέλο. Εγώ πλέον, εγώ ο ίδιος, μέσω του ίντερνετ κλείνω τις διακοπές μου. Το ίδιο κάνουν και οι περισσότεροι συμπατριώτες μου στην Ευρώπη 23% των ταξιδιωτών οργανώνουν μόνοι τους τα ταξίδια τους. Σε κάποιες χώρες όπως τη Σουηδία ε, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει πάνω από το 40%. Οι ταξιδιώτες που αγοράζουν στο ίντερνετ, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, δεν γνωρίζουν ότι η προστασία των συμφερόντων τους μέσω του ίντερνετ είναι πολύ μικρότερη από ότι αν προχωρήσεις μέσω ενός ε, ε, πρακτορείου. Είναι θετικό λοιπόν το ότι θέτει το θέμα αυτό η Επιτροπή. όντω τα 20 χρόνια παρά είναι μεγάλη χρονική περίοδο. Ελπίζω να μπορέσει η Επιτροπή σήμερα να μας πει πότε θα αναθεωρηθεί η οδηγία και ποιε θα είναι οι αλλαγέ στο κείμενο. Δεν θα πρέπει να μιλούμε στο Ευρωπαϊκό Νογιούλο υπέρ του ηλεκτρονικού εμπορίου, να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό το e-commerce και διασυνοριακά και να μην μπορούμε να προσφέρουμε τις βασικές, ε, τη βασική προστασία σε αυτούς. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό κύριε Μόλτσερ. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν μοναχά διαφορές ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών, αλλά και στην, στον ορισμό των ε, οργανωμένων ταξιδίων που δημιουργούν προβλήματα. Το να υπάρχει μια ενιαία βάση και κοινή κανόνες παιχνιδιού είναι κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 15 χρόνια. Η αναθεώρηση αυτής της γενικής βάσης είναι απαραίτητη όμως για να εξασφαλίσει την ενότητα και την ελευθερία κυκλοφορία σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ δεν νομίζω ότι η σωστή αντιμετώπιση είναι να υπάρξει απόλυτη ισοπαίδωση και εξίσωση σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι μια τέτοια ισοπαίδωση και απόλυτη ομοιόμορφη αντιμετώπιση θα έχει πολύ σοβαρές δυσκολίες για τα γραφεία ταξίδιων. Θα πρέπει εμείς καταρχήν να δώσουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο καταναλωτής το ίντερνετ αλλά με ανάλογη υπευθυνοποίηση των γραφείων ε, ε, ταξίδιων. Σαν παράδειγμα το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές φορές πληροφορίες παραπλανητικές όπως αυτές που αφορούσαν τις πρόσφατες απεργίες στην Ελλάδα και οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν την ε, εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Για την περίπτωση της Ελλάδος φοβάμαι ότι θα υπάρχουν και περαιτέρω απεργίε. Εμεί ελπίζω ότι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ο κρατικό μηχανισμό στη χώρα αυτή και να διατηρηθεί η προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ο Κόζα. Για δύο λεπτά. Κυρία Κόζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής θέμα. Ο κύριος Κάλλας, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, όταν ήταν στη διαδικασία ακρόαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε τονίσει μια αξία η οποία κατά την άποψή του ήταν προεξάρχουσα. Δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια απόλυτη διατήρηση των δικαιωμάτων του κάθε ατόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως απαιτεί να υπάρξει μια συνένωση και μια ε, εν, ε, όλων, ενοποίηση μάλλον όλων των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών για την, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα ενιαίο χάρτη. Η Ισπανική Προεδρία και τονίσει ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να είναι κομμάτι της Προεδρίας σας. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το θέμα αυτό, γιατί η οδηγία η οποία ήδη έχει ηλικία 20 ετών, λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα πολλών καταναλωτών, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη πολλές φορές τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες ούτε σε μεμονωμένα ταξίδια, ούτε σε ταξίδια τα οποία είναι οργανωμένα. Επομένως, εγώ τονίζω την ανάγκη να υπάρξει μια χάρτα δικαιωμάτων των ταξιδιωτών η οποία να έχει ενιαίο χαρακτήρα και η οποία θα παρέχει και τι απαραίτητε εγγύησει για τα άτομα με αναπηρίε και προβλήματα και η οποία θα καλύπτει τι ανάγκε των ατόμων αυτών ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια. Αν επιτευχθεί λοιπόν κάτι τέτοιο να υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση τότε μονάχα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πραγματικά ελευθερία διακίνηση όλων των ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τικάου για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια καλύπτει θέματα και μεταφορών και άλλων υπηρεσιών που αφορούν και θέματα δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς και άλλων προμηθευτών τουριστικών υπηρεσιών. Η οδηγία του 90 δεν λάμβανε υπόψη της πρόσφατες εξελίξεις όπως τις κρατήσεις τουριστικών υπηρεσιών από το ίντερνετ. Το 23% του ευρωπαϊκού τουρισμού και μεγάλο ποσοστό επίσης των νοικοκυριών ταξιδεύει μέσω ίντερνετ, οργανώνει τα ταξίδια του μέσω ιστοτόπων. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί η οδηγία για να συμπεριλαμβάνει και όσους ε, προσφέρουν αυτές τις δυναμικές υπηρεσίες έτσι ώστε οι καταναλωτές και οι καταναλώτριες να έχουν εγγύηση των δικαιωμάτων τους για κάθε προσφορά που βλέπουν στο ίντερνετ. Επίσης νομίζω ότι οι σελίδες που προσφέρουν τέτοιες τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να τυχαίνουν κάποια εγγύηση ή πιστοποίηση για να είμαστε βέβαιοι για την ταυτότητά τους τουλάχιστον και να υπάρχει μία εγγύηση χορήγησης πληροφοριών. Μια μελέτη του 2009 που έκανε η Κομισιόν σε σχέση με τα οργανωμένα ταξίδια, τα δυναμικά αυτά οργανωμένα ταξίδια από το Ιντερνετ δηλαδή, έδειξε ότι το ποσοστό των ηλεκτρονικών κλεισμένων ταξιδίων έχει ανεβεί στο κατά 12% από το σύνολο του 28. 66% δε είναι άμεσες πληρωμές από το, την ιστοσελίδα ή κρατήσεις της τελευταίας στιγμής από ειδικέ σελίδε της τελευταία στιγμή. Αυτό το προτιμούν οι καταναλωτές γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα, χαμηλότερες τιμές σε σχέση με, τις, με τα παραδοσιακά πρακτορία ή γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους παραδοσιακά πρακτορία. Οι πληρωμές για τα οργανωμένα αυτά ταξίδια καμιά φορά μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να γίνουν. 70% των παραπώνων που ελήφθησαν πέρυσι από ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων δικαιωμάτων των καταναλωτών και καταναλωτριών αφορούσαν αυτά τα οργανωμένα ταξίδια και λανθασμένες πληροφορίες πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή αφορούσαν χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών ή χαμηλότερη απόση έγγραφε στις διαφημίσεις. Πρέπει λοιπόν, είναι καιρός να αναθεωρηθεί η οδηγία κύριος εγραφε στι διαφημισει πρεπει λοιπον ειναι καιρο να αναθεωρηθει η οδηγια αυτη ευχαριστουμε ο Χάρμπορ. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, θα ευχαριστήσω τον Επίτροπο και από την ομάδα μου και ως πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Ε, ήταν πολύ επίκαιρη η παρουσία του σήμερα. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί απάντησε πάρα πολύ γρήγορα στην προφορική ερώτηση τη Επιτροπή μου τη 3η Δεκεμβρίου που έθεσε μια σειρά θεμάτων και στην οποία απάντησε συνολικά και πλήρω. Πιστεύω ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μα όπως ε, καθώς προετοιμάζει τις θέσεις της Επιτροπής ώστε και η δική μου Επιτροπή και η Επιτροπή Μεταφορών να συζητήσουν και να εξετάσουν από κοινού πολλά από τα θέματα που τέθηκαν για την πρόταση αναθεωρήσης οδηγίας δεδομένης της φύσης και των αλλαγών ε, στον χώρο των οργανωμένων ταξιδίων, θέμα που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι σήμερα, η νέα οδηγία θα πρέπει να είναι ασφαλής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να είναι άκαμπτη όταν προσπαθεί να προεξοφλήσει τις ε, μελλοντικέ ανάγκες των ανθρώπων. Πιστεύω ωστόσο ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε, και το λέω στην Επιτροπή, είναι ότι υπάρχουν και άλλες διαστάσεις που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για την προστασία των καταναλωτών θέματα ασφάλειας των ξενοδοχείων. Με μικρά παιδιά υπάρχει ασφάλεια στην πισίνα. Ε, η προστασία από τις πυρκαγιές. Χρειάζεται να υπάρχουν σωστοί δείκτες, ε, σωστή σήμανση ε, που μπορεί να γίνει με αθελούσια συμφωνία, αλλά πιστεύω ότι η πρόταση πρέπει να είναι και εκτεταμένη και φιλόδοξη. Πιστεύω ότι αυτό θέλετε να κάνετε και θα σας υποστηρίξουμε πλήρως την παρουσίαση μιας τέτοιας πρότασης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι μας θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πιο απτό και συγκεκριμένο χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι θα δίνει την απαραίτητη προστασία για τα εκατομμύρια ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ταξιδεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με οργανωμένα ταξίδια, ιδίω για πακέτα διακοπών χρειαζόμαστε να έχουμε μια σωστή παρέμβαση ώστε να μπορέσει η αρμόδια οδηγία να επικαιροποιηθεί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές από ένα φυλάδιο, από ένα προσπέκτους αποφασίζουν να, να αγοράσουν ένα ταξιδιωτικό πακέτο, αλλά συγχρόνως είναι πολύ περισσότεροι οι καταναλωτές οι οποίοι χρησιμοποιούν το ίντερνετ για την κράτηση ταξιδίων και έχουμε μια ανάδυση νέων φαινομένων όπως είναι οι εταιρείε χαμηλού κόστους και επίσης η χρήση κρουαζιεροπλοίων για οργανωμένες διακοπές. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ε, μιας επανεπεξεργασίας αρμόδιας οδηγίας. Καταρχήν να δούμε τι ακριβώς καλύπτει ο τομέας των οργανωμένων ταξιδιών και στη συνέχεια να δούμε πού βρίσκεται η αστική ευθύνη των φορέων των ταξιδιωτικών, ώστε να υπάρξει η απαραίτητη και λογική ε, υποστήριξη των καταναλωτών σε περίπτωση χρεοκοπίας πτώχευσης των επιχειρήσεων που παρέχουν τις ταξιδιωτικές αυτές υπηρεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο λοιπόν για την καλή προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Ο κ. Κάζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την πρόταση του νέου Επιτροπή. Ακούσαμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση στη, υπήρξε αύξηση στην αγορά των ε, ταξιδίων, των ταξιδίων από ίντερνετ που προσφέρουν πολύ μικρότερη προστασία σε σχέση με την αγορά ενός ε, ταξιδιωτικού πακέτου που παρέχεται από ένα πρακτορείο αλλά το κόστος ε, ε, οι αγορές μάλλον από τη, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία έχουν μια προστιθέμενη αξία ακριβώς για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της οδηγίας. Η οδηγία έτσι δεν προστατεύει παρκώς τον καταναλωτή και δημιουργεί μια ανισορροπία στην τουριστική βιομηχανία. Θα ζητούσαμε λοιπόν από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ισότιμη μεταχείριση, ισότιμη αντιμετώπιση όλων των καταναλωτών άσχετα από το που αγοράζουν το πακέτο. Η προστασία του καταναλωτή πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας και θεωρώ, πιστεύω ότι και η Επιτροπή αυτό, σε αυτό στοχεύει. Ωστόσο πιστεύω ότι η ορολογία, οι ορισμοί θα πρέπει να ενημερωθούν, να γίνουν πιο επίκαιροι να, σε ό,τι αφορά την έννοια του καταναλωτή, του πολιτή, του, του operator, αλλά και η εμβέλεια η ίδια της οδηγίας πρέπει να επεκταθεί. Κατά την άποψή μου, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ε, τηρεί τις διατάξεις της οδηγίας αν από το πώς πωλείται το πακέτο, ε, ανεξάρτητα ή μέσω πρακτορείου. Ο επιχειρηματίας, ο τελικός επιχειρηματίας είναι ένας επιχειρηματίας που πωλεί μία υπηρεσία με το όνομά του Προσφέροντα ταυτόχρονα πρόσβαση στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει το πακέτο. Πιστεύω ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα δουλέψει και ο Επίτροπος. Ελπίζουμε ότι τα δικαιώματα του καναλωτή θα προστατευτούν καλύτερα. Κυρία Σεναλόβα, δύο λεπτά. Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, η αναθεώρηση τις οδηγίες για τα οργανωμένα ταξίδια αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση στον τομέα του τουρισμού που συνδέεται πολύ με τις νέες τεχνολογίες και την εξέλιξή τους αλλά και τις εξελίξεις στον τομέα της πώληση υπηρεσιών. Εγώ θα μιλήσω μόνο για την πώληση μέσω ίντερνετ που εξελίχθηκε σημαντικά από την αύξηση του, των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους. Ε, προφανώς όλα αυτά προσφέρουν ευκολίες πρόσβαση αλλά και απειλές ταυτόχρονα για την προστασία του καταναλωτή. Πριν από λίγους μήνες η Επιτροπή Μεταφορών έθεσε μια ερώτηση στην Επιτροπή που αφορούσε ε, μια ε, εταιρεία χαμηλού κόστους που πτώχευσε. Ε, την εποχή εκείνη οι ταξιδιώτες έμειναν στα αεροδρόμια χωρίς κανένα μέσο επιτροπή επιστροφή, ή με πολύ δύσκολο μέσο επιστροφή, τότε διαπιστώθηκε πραγματικά η με πολυ δυσκολο μεσο επιστροφή. τοτε διαπιστωθηκε πραγματικα η ανεπαρκη προστασια των ε, ταξιδιωτών. Ε, πρέπει η Επιτροπή να, αντιμε... να βρει τρόπου για να αντιμετωπίσει τέτοιε καταστάσει προ όφελο των καταναλωτών. Σε λίγου μήνε ξεκινούν οι καλοκαιρινέ διακοπέ. Δεν θέλουμε να επανέλθει το πρόβλημα όπως αυτό που είχαμε πέρσι με την πτώχευση του, του Sky Europe. Ε, τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν βάσει ενός κοινού παρονομαστή προστασία του καταναλωτή με καλύτερη ενημέρωσή του για τους όρους και την τιμή των υπηρεσιών. Μια τελευταία παρατήρηση για την δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε η Επιτροπή. Κατά την άποψή μου είναι αναγκαίο να επιτρέψουμε να να γίνουν οι διαβούλευσεις αυτές σε όλες τι επίσημε γλώσσε στην Ένωση, σαν θέλουμε να έχουμε την άποψη όλων ε, για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Διότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν το ίδιο δικαίωμα στην ενημέρωση και το ίδιο δικαίωμα στο να παρέχουν την άποψή τους για την ενημέρωση. Η κυρία Φώστερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω το τρίτο σημείο της προφορικής ερώτησης για την περίπτωση πτώχευσης αεροπορικών εταιριών. Ένα ψήφισμά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είχε ζητήσει να υπάρξει ένα ειδικό ταμείο για την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας αλλά φυσικά θα πρέπει ο ίδιος ο καταναλωτής να χρηματοδοτεί αυτό το ταμείο, δηλαδή αυτό θα αύξανε το κόστος των εισιτήριων. Αυτό θα πρόσθεται όμως στο ίδιο επαχθές βάρος των αεροπορικών φόρων, των φόρων αεροδρομίου και όλων αυτών των πρόσθετων τελών που πρέπει να καλύψει ο καταναλωτής. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται σε εθνικό επίπεδο οι απαραίτητε υποχρεώσει των ρυθμιστικών αρχών για την πολιτική αεροπορία, όπω είναι ο έλεγχο των ισολογισμών των εταιριών και οι σωστέ διαδικασίε σε περίπτωση εκαθάριση εταιριών. Θέλουμε λοιπόν η Κομισιόν να το πράξει αυτό και επίση έχουμε ζητήσει από την Κομισιόν να εξετάσει άλλε δυνατότητε για την αποζημίωση των επιβατών σε αυτήν την περίπτωση και επίση την παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών σε σχέση με την ασφάλεια, με τους κινδύνους και όλα αυτά τα συστήματα. Ο κύριο Higgins για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι επικροτήσαμε την αναγγελία στις 29 Αυγούστου του 9 από τον πρώην Επίτροπο ότι η παρούσα οδηγία είναι τελείως επιχειωμένη και δεν καλύπτει τις προκλήσεις και τις ανάγκες των οργανωμένων ταξιδίων σήμερα αλλά και και των πελατών πολλοί λόγοι αναφέρθηκαν ε, σήμερα. Η οδηγία ήταν καλή στο παρελθόν, τώρα ωστόσο δεν έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις των ταξιδιωτών. Δεν εξετάζει και δεν λέμε υπόψη την, ή ε, αύξη, την αυξανόμενη τάση αγοράς ε, των ε, ταξιδιωτικών προϊόντων από τους ίδιους τους καταναλωτές ή από τις αγορές εκτός επικράτειας. Όλο και περισσότεροι πολίτες σήμερα οργανώνουν μόνοι τους τα πακέτα διακοπών τους μέσω της εύκολης πρόσβασης που έχουν στο ίντερνετ, στο παρελθόν ε, το ποσοστό των ταξιδιωτών που προστατεύονται έπεσε από το 90% στο 60% περίπου. Άρα τα υφιστάμενα μέτρα δεν καλύπτουν μια σειρά ε, περιπτώσεων αγοράς από online ή ε, από εκτός, εκτός χώρας προγραμμένων ταξιδιών όντως στην Ένωση έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν πετύχει πολλά πράγματα για τον καταναλωτή. Αν δούμε όμω την παρούσα κατάσταση για τα οργανωμένα ταξίδια και την προστασία των ταξιδιωτών θα δείτε, θα συμφωνήσουμε ότι η Ένωση είναι πιο λιγότερο ενοποιημένη αγορά από οποιαδήποτε άλλη εμπορική, από οποιοδήποτε άλλο εμπορικό μπλοκ. Και υπάρχει σύγχυση για το ποιο έχει την ευθύνη, ποιο καλύπτει τα κενά και το κόστος, τι γίνεται με την παλιότερα. Υπήρχε προστιθέμενη προστασία αν αγόραζες μέσω ε, με, με πιστοτική κάρτα. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Στην επιπλέον έχουν υπάρξει μία ε, σύγχυση μεταξύ αεροπορικών εταιριών, πρακτορείων τουρισμού, πρακτορείων κουραζιερών κλπ. Χρειάζεται λοιπόν μία πολύ εξελιγμένη ε, οδηγία που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες τεχνολογίες για να λάβει ε, υπόψη τις αλλαγές, να διευκρινίσει την κατάσταση και να προστατεύει καλύτερα τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούρκης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Υποστηρίζω την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, αλλά με έχει απογοητεύσει. Δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, όπου πάνω των 50% των ταξιδιωτών αυτοοργανώνονται και χρησιμοποιούν χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά το εύρος της πρέπει να καθοριστεί σαφώς. Δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να αγνοείται τι ακριβώς καλύπτει. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Δεν είναι σωστό να επεκτείνεται το εύρος της για να καλύπτεται και τις λεγόμενες δυναμικές εταιρείε οργάνωση ταξιδίων διότι αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθεί το κόστος του ταξιδιού για τον, για τον ταξιδιώτη. Αν κανείς κάνει μια κράτηση ξενοδοχείου αμέσως μετά την κράτηση του αεροπορικού εισιτηρίου και θεωρηθούν όλα αυτά σαν ένα σύνολο δεν πρέπει να αφήσουμε τον καταναλωτή μόνο του έρημο γιατί κανείς δεν μπορεί να καλύψει και τα δύο ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε η κυρία Ράνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το σημαντικό ρόλο που παίζει η τουριστική βιομηχανία στις χώρες μας. Σχεδόν ο καθένας από εμά έχει σχέση με κάποιο τομέα της τουριστικής βιομηχανίας. Και επομένως για τις χώρες μας έχει μια μεγάλη σημασία αυτό το ερώτημα και χαίρομαι που ο Επίτροπος ο κ. Σταλή έχει ήδη επιληφθεί του θέματος αυτού στην αρχή της νέας Κομισιόν. Η ελευθερία διακίνησης, η ελευθερία ταξιδίων είναι μια ελευθερία η οποία έχει πάρει ένα άλλο ποιοτικό χαρακτήρα λόγω της ποσοτικής αλλαγή στον αριθμό των ατόμων οι οποίοι ταξιδεύουν. Πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Χάρη στο ίντερνετ έχει υπάρξει και τροποποίηση στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στον τρόπο με τον οποίο κλείνουν ταξίδια αλλά ιδίω επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή οικονομική κρίση, είναι απαραίτητο εμεί να κάνουμε τι απαραίτητε προσπάθειε για να προστατεύσουμε του πολίτε μα. Να μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή τη ελευθερία διακίνηση. Είναι λοιπόν απαραίτητο όταν χρησιμοποιούν τις οικονομίες τους που πολλές φορές έχουν με μεγάλο κόπο αποκτήσει για ταξίδια να έχουν την πλήρη αυτή προστασία. Δεν πρέπει το γεγονός ότι είναι φτηνότερες πλέον οι πτήσεις και οι προσφορές από το ίντερνετ να υπονομεύσει τα δικαιώματά τους. Ένα ερώτημα ακόμα το οποίο θα ήθελα να υποβάλω στον κύριο Επίτροπο. Ποιες είναι και οι εγγυήσει οι οποίες υπάρχουν για τους ε, επιβάτες των αεροπορικών εταιριών. Ξέρουμε ότι οι αεροπορικέ εταιρείε κινδυνεύουν όλο και περισσότερο να πτωχεύσουν όταν τα χρέη του σωρεύονται συνέχεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα μπορέσει το ταχύτερο δυνατό να μα υποβάλει μια πρόταση η οποία θα λάβει υπόψη το πρόβλημα αυτό τη ε, μη φερεγγιότητα των ε, αεροπορικών εταιριών και το οποίο είναι σημαντικό για να καλυφθούν και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών που πηγαίνουν διακοπές. Ευχαριστώ. Κύριος Παπα-Νικολάου, στη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, στην εποχή μα η ευρεία χρήση του διαδικτύου επιτρέπει στου καταναλωτέ να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζουν ακόμη και τι διακοπέ του, να του δίνεται δηλαδή η δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να μην αγοράζουν έτοιμα πακέτα όπω είχαμε μάθει μέχρι τώρα, αλλά να επιλέγουν μόνοι του πώ θέλουν να οργανώσουν τι διακοπέ του. Και βεβαίω με την εμπλοκή περισσότερων παραγόντων πλέον τίθεται το ερώτημα ποιο είναι ο υπεύθυνο σε περίπτωση πλημελού εκπλήρωσης παροχή και βεβαίω από ποιον θα ζητήσει τελικά ευθύνη ο καταναλωτής. πολύ σωστά αναφέρθηκε και από του συναδέλφου και πρέπει να δώσουμε απαντήσει να εξυγχρονίσουμε την οδηγία την οποία έχουμε μέχρι σήμερα. είναι καθοριστικό και για την ελλάδα αυτό που όπω γνωρίζετε είναι τουριστικό προορισμό και όσο πιο ξεκάθαρα ορίσουμε ποιο είναι κάθε φορά ο υπεύθυνο ο έλληνα ξενοδόχο το ε, τουριστικό πρακτορείο οποιοδήποτε εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή τόσο πιο αξιόπιστοι θα είναι όλοι εκείνοι που αναπτύσσουν ε, δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού. θέλω να κλείσω λέγοντα ότι η νομική προστασία των ευρωπαίων πολιτών είναι καθοριστική παράλληλα όμω είναι ευθύνη κύριε επίτροπε να ενημερώσουμε για τα δικαιώματα που μέχρι σήμερα έχουν όλοι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν διακοπέ σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα Κυρίω όμω να του ενημερώσουμε για τα κενά και για τι βελτιώσει που θέλουμε να κάνουμε. είναι σημαντικά όλα αυτά να το μάθουν όμω και οι πολίτε για να αξιοποιούν αυτά του τα δικαιώματα. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Το κύριε Πρόεδρε, τα περισσότερα έχουν υποθεί. Θέλω όμως να εστιάσω σε τέσσερα σημεία. Η οδηγία αυτή είναι 20 χρονών. Για κορίτσι τα είκοσι χρόνια είναι μια πολύ καλή ηλικία. για οδηγία τα είκοσι χρόνια σημαίνουν ότι χρειάζεται η οδηγία lifting και αυτό γιατί μπήκαν τέσσερα πράγματα στη ζωή μας. το ένα είναι το ίντερνετ. καθώς μπήκε το ίντερνετ στη ζωή μας μπορούμε να διαλέξουμε τις διακοπές μας στο πιο απομακρυσμένο μέρος του κόσμου χωρίς να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. όταν θα πάμε εκεί όμως ίσως να διαπιστώσουμε ότι θα έπρεπε να το είχαμε ξανασκεφτεί. το δεύτερο είναι οι τιμές. ο καταναλωτής έχει υποχρέωση αλλά έχει και δικαίωμα να ξέρει αν οι τιμές ανάμεσα στις οποίες καλείται να διαλέξει βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητος αν δηλαδή δεν υπάρχει αφέμητος ανταγωνισμός. το τρίτο είναι η ποιότητα ένα κατάλημα που σε ένα κράτος μέλος μπορεί να θεωρείται εξαιρετικό από έναν πολίτη άλλου κράτους μέλους μπορεί να θεωρείται μέτριο. και τέλος υπάρχει το θέμα της ασφάλειας. επειδή οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι που μαζεύουν με πολύ κόπο τα χρήματα για να κάνουν διακοπές πρέπει οφείλουμε να τους κάνουμε να νιώθουν ασφάλεια. αυτά ζητούμε από τη νέα οδηγία. Πάντως, θα σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Σον Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, πολλοί συνάδελφοι τόνισαν την ανάγκη του να υπάρξει αυτή η αναθεώρηση της ε, αρμόδιας οδηγίας, το ταχύτερο το καλύτερο. Και φυσικά έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή. Επειδή όμω η οδηγία αυτή πρέπει να ευνοήσει τον καταναλωτή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πλήξει την τουριστική βιομηχανία. Μπορεί να βοηθήσει και τη βιομηχανία και τον καταναλωτή. Εγώ έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή το γεγονό ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουμε δύο εκατομμύρια άτομα τα οποία θα περάσουν τα 60 του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία στην τουριστική βιομηχανία να εκμεταλλευτεί την δυνατότητα ταξιδίων αυτών των ατόμων χωρίς να του δημιουργεί προβλήματα. Και εδώ πρόκειται για ταξίδια περιεκτικά που καλύπτουν όλες τις πτυχές των ταξιδιών. Πρέπει λοιπόν να αντλήσει το δυναμικό των υπερεξικοντούτιδων η βιομηχανία, η τουριστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και η οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση, θα πρέπει να θεωρηθεί αυτή η οδηγία σαν μια ε, θετικού αθροίσματος πρόταση και για τον καταναλωτή και για την τουριστική βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κάλτεμπάχα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Έχουμε μητέρα μεγάλης οικογένειας και έχω μάθει τα τελευταία χρόνια να διαβάζω καταλόγους, φυλάδια για μεγάλα ταξίδια που είναι δύσκολο να τα καταλάβουν ακόμα και οι εργαζόμενοι στα τουριστικά γραφεία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εγώ να παρουσιάσω την άποψή μου ως καταναλώτρια σε σχέση με την οδηγία και να τονίσω τη σημασία να υπάρχει δυνατότητα συγκρισιμότητας μεταξύ των φυλαδιών και των προτάσεων ώστε να μπορέσει να επιλέξει ο καταναλωτής. Πολλές ε, προσφορές έχουν ε, ε, προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν παιδιά μέχρι 6 ετών, άλλες 10 ετών, Όλε άλλε λένε ότι το πρώτο παιδί έχει μια έκπτωση α, το δεύτερο παιδί έχει μια έκπτωση β. Διαφορετική, χαμηλότερη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μια σαφήνεια σε όλα αυτά τα πράγματα για να υπάρχει και η κατάλληλη προστασία των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει μια σωστή αλλά συγκρίσιμη πληροφορία προ τον καταναλωτή για να μπορεί να πράγματι να επιλέξει. Σα ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Στήλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Επίτροπο να υποστήριξω και εγώ τους συναδέλφους που είπαν ότι πρέπει να προστατεύσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες ε, ε, ταξιδιωτών, τη γίνεται στα ξενοδοχεία, με την προστασία των παιδιών, με την προστασία από την πυρκαγιά. Είδαμε στο παρελθόν μια σειρά προβλημάτων. Δύο συγκεκριμένα θέματα ωστόσο θέλω να θίξω. Ακούσαμε το ενδεχόμενο ε, ε, προμηθειών από πιστοποιητικέ τράπεζε. Όλο και περισσότερο κόσμο χρησιμοποιεί πιστοποιητικέ ε, κάρτε, θεωρώντα ότι έχει προστασία μέσω αυτών. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι ευρωπαϊκέ εταιρείε, επιβαρύνοντα τι πιστοποιητικέ κάρτε ή περνώντα περισσότερες από μία φορές ε, ε, επιβάλλοντας προμήθειες έστω και αν έχεις ε, προ, προ, παίρνει ένα εισιτήριο για τέσσερα άτομα, σε χρεώνουν τέσσερις φορές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν, δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα αποσμίωσης γιατί σε πολλές οικογένειες αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα όταν επιλέγουν τις διακοπές τους. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, τα 20 τελευταία χρόνια η αγορά ταξιδιών αναπτύχθηκε δυναμικά. Πολλοί κόσμος αγοράζει πλέον μόνο του τα ταξίδια. Οι φυστάμενες διατάξεις του οδηγίας ωστόσο δεν εφαρμόζονται σε τέτοια ε, δυναμικά πακέτα ταξιδιών που σημαίνει ότι ο κόσμος ταξιδεύει χωρίς προστασία θα πρέπει να δώσουμε σαφέστερο περιεχόμενο στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, προστατεύοντα περισσότερου ταξιδιώτε. Επίση, πρέπει να ορίσουμε καλύτερα την έννοια τη ευθύνη σε περίπτωση ε, πτωχεύσεω ε, επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, με, σε πάρα πολλέ περιπτώσει πτωχεύσεων, ο, οι ταξιδιώτε έμειναν, έμειναν στα αεροδρόμια. Χρειάζεται λοιπόν να αναθεωρήσει οδηγίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει τη διαδικασία Catch the Eye και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αρμόδιο κύριο Επίτροπο Ντάλι. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις απόψεις των εντύμων. Άκουσα την απόψη όλων των εντύμων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σημαντικό το ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει για την οδηγία αυτή. Ορισμένοι έχουν υποστηρίξει την προσέγγιση της Κομισιόν, αλλά έχουν υπογραμμίσει διάφορες επιμέρους πτυχές της προτινόμενης οδηγίας και τα έχω καταγράψει όλα αυτά και θα λυθούν όλα αυτά υπόψη στις συζητήσεις και τις διαβολεύσεις που θα ακολουθήσουν για τη μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας. Θέλω να σας διαβου... βεβαιώσω ότι η Κομισιόν λαμβάνει πάρα πολύ στα σοβαρά όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχετε εγείρει και είναι έτοιμη να διερευνήσει τις καλύτερε δυνατέ λύσει για την αναθεωρημένη οδηγία. Βρισκόμαστε στο μέσο τη διαδικασία. Διαβούλευση. Αναλύουμε την ανάδραση που έχουμε πάρει από το κοινό, από τους καταναλωτές, από τις οργανώσεις επιχειρήσεων, αλλά και από τα κράτη-μέλη που έχουν όλοι οι φορείς αυτοί συμβάλει στην ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης. Μπορώ επίσης να σας πω ότι θα οργανώσει ένα ατελιέ για τους εμπλεκομένους τον Απρίλιο του 2010 η Κομισιόν, που θα εστιάσει την προσοχή του στις δυνατότητες επιλογών για την αναθεώρηση του πακέτου αυτού τις οδηγίες μάλλον για τα ταξιδιωτικά πακέτα και θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν στην συζήτησή μας. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε την κατεύθυνση που θα λάβει η οδηγία αυτή προτού τελειώσει η διαδικασία αντιμετώπισης του αντικτύπου και της διαβούλευσης, αλλά σίγουρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο στόχος μας είναι